Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε νομίζω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Είναι η τελευταία ημέρα και βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που εγκαταλείπουν τις Βρυξέλλες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να μην πέσουν στην κίνηση. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στη μέση διάταξη να πάμε στο σημείο 12 αφού ακούσουμε ένα μήνυμα από τους διερμηνείς Βρισκόμαστε στη 38η μέρα των κινητοποίησεών μας ε, κατά της επιβολής ε, από το Γενικό Γραμματέα Συνθηκών Εργασίας που δεν εγγυώνται την ποιότητα της δουλειάς μας. Ε, ως εκ τούτου δεν θα παραχωρήσουμε υπέρβαση ωραρίου, λυπούμεθα γι' αυτό. Έχουμε δει κάποια πρόοδο ε, σε ό,τι αφορά ε, τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, στην Ποσαχάρη, Αφρική, η ποιότητα έχει βελτιωθεί 87% ε, των παιδιών βέβαια εξακολουθούν να μην έχουν κατάλληλο επίπεδο αλφαβετισμού. Μέχρι το 2030 χρειάζονται 89 εκατομμύρια ε, δολάρια ε, που πρέπει να επενδύονται κάθε χρόνο στην εκπαίδευση. Και αυτή τη στιγμή 16 δις στην εκπαίδευση είναι το ποσό. Καταλαβαίνετε τόσο το μέγεθος της πρόκλησης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί το 20% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας να τα δώσει για κοινωνική ένταξη, ανθρώπινη εξέλιξη και μεταξύ αυτών εντάσσεται παιδεία και υγεία. Ο εισηγητή μα ε, για το σημείο 12, λοιπόν, αναπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη εκπαίδευση, είναι ο κύριο Βίνσεντ Πεγιόν. Θα μα πει περισσότερα. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει μείωση των κονδυλίων για την Αφρική ιδίω. Ε, μα ενδιαφέρει το πρόβλημα λόγω τη έλλειψη εκπαίδευση για τα παιδιά και του νέου. Φυσικά, ένα άλλο θέμα είναι η προσφορά θέσεων εργασία. Και αυτό ήταν και το θέμα τη συνόδου του Αμπιτζάν και Γνωρίζω από την εμπειρία μου ε, τι γίνεται στην Αφρική και σε κάποιες γειτονικέ χώρες. Η ποιότητα της εκπαίδευσης, ο αριθμός των παιδιών στο σχολείο που είναι πολύ μικρό καθιστά πάρα πολύ δύσκολο ε, την ε, ε, παροχή βοήθειας και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση και τις στόχες. Η έκθεση του κυρίου Παγιό είναι πάρα πολύ καλή. είναι η τελευταία έκθεση του Κοινοβουλίου σε αυτή τη θητεία που πρέπει όμως να δώσει κάποια σημεία αναφοράς για το επόμενο Κοινοβούλιο. δεν ξέρω αν Υπάρχει κάποιο άλλο να δώσει το λόγο στον Βενσάν Πεγιό. Ευθύ αμέσω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι είμαστε ακριβώς ε, λίγες μέρες πρώτων ε, διακοπών. Ε, μου ζητήσατε να σας παρουσιάσω νωρίτερα την έκθεση, αληθεύει αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα για προσωπικούς λόγους να είμαι νωρίτερα εδώ. Είπατε εσείς τα ουσιώδη, πάρα πολύ γρήγορα και εγώ, να πω ότι αυτή η έκθεση κατά την άποψή μου ήταν απαραίτητη, ήταν αναγκαία διότι η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που περιορίζεται στην εκπαίδευση, έχει να κάνει με τη δημοκρατία, την οικονομική ανάπτυξη, την ίδια την ασφάλεια και πολλές φορές η εκπαίδευση για όλου αυτούς του τομεί παίζει μείζωνα ρόλο, η εκπαίδευση των παιδιών, των μαθητών, των πολιτών εν γέννη. Αλλά Υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο. Στην πραγματικότητα, παρότι υπάρχουν αλλαγές από το 2016 και μετά, η αναπτυξιακή βοήθεια για την εκπαίδευση μειώθηκε σημαντικά. Αυτό δεν είναι γνωστό ε, στη δεκαετία πριν το 2016. Υπάρχει δηλαδή ανάγκη να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος που δεν έχει όμως καλυφθεί επαρκώς ακόμη. Το είπατε και εσείς ε, Υπάρχει κάποιο είδους υποκρισία, υπάρχει ένα παράδοξο, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Στόχος 4, στο πλαίσιο των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει λοιπόν να ε, εξαπλασιαστεί ουσιαστικά η αναπτυξιακή βοήθεια σε σχέση με το τι προβλέπεται μέχρι το 2030. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, προσπαθούμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ λόγων και έργων. Αναλαμβάνουμε δε, με, ε, παίρνουμε μεγάλο κίνδυνο, για την Αφρική όπως είπατε, γιατί δεν διαθέτουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Και, και περιμένω ε, ε, και πώ θα ολοκληρωθούν οι συνομιλίε με την Κομισιόν, αλλά είναι θετικέ οι συνομιλίε μέχρι τώρα. Στην τελευταία τη ανακοίνωση η Κομισιόν την εκπαίδευση, μάλλον η τελευταία τη ανακοίνωση είναι από το 2002. Και πρέπει λοιπόν να, να δοθεί μια νέα όθηση. Ε, το 2010 είχαμε ένα έγγραφο εργασία ε, που επικαιροποιεί την κατάσταση, αλλά η τελευταία ανακοίνωση για την εκπαίδευση, όπω είπα, είναι από το 2002. Δεν έχουν περάσει 16 χρόνια. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ ε, το χρονικό αυτό διάστημα και έχουν γίνει έκτοτε διάφορα. Ο στόχο είναι πολύ απλό και θέλω να εργαστώ ως εξή. Να καταθέσω μια έκθεση που θα αναφέρει κάποια βασικά σημεία ε, που θα τα στηρίξει πιστεύω η, ομο... η πλειοψηφία τουλάχιστον για να μην πω το σύνολο των συναδέλφων βουλευτών ώστε το μήνυμά μας να γίνει ακουστό δεν χρειάζεται να βάλουμε λεπτομέρειες ε, πάνω στις λεπτομέρειες και να λεπτολογούμε τα πράγματα. Απλά κάποιες βασικές γραμμές να ε, προβάλλουμε. Ε, είναι λίγο διαφορετική η μέθοδος από ό,τι κατά το παρελθόν. Πριν τις συζητήσεις για τις τροπολογίες είχα συναντήσεις με τους σκιώδεις συζητητέ από τις άλλες πολιτικές ομάδες, ώστε από κοινού να καταρτήσουμε τις προτεραιότητές μας με κοινή συμφωνία. Είπα και Επαναλαμβάνω, ξέρετε ότι δεν είναι η πρώτη μου θητεία ως Ευρωβουλευτό, αλλά δεν θεωρώ ότι όσο περισσότερες λεπτομέρειες έχει το κείμενο γίνεται καλύτερο, αντίθετα νομίζω αλλοιώνεται. Και με τις ε, τροπολογίες ε, πολλές φορές ε, όταν βάζουν πάρα πολλές τροπολογίες χάνει το κείμενο την αρχική το αρχιτεκτονική αλλοιώνεται γι' αυτό λοιπόν θέλω να το περιορίσουμε Τώρα, πρώτη βασική ιδέα. Η εκπαίδευση, πολύ απλή ιδέα, πρέπει να ξαναμπεί στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε δείκτες πολύ πιο συγκεκριμένους για την εκπαίδευση, άρα να μην εμπλέξουμε την εκπαίδευση με τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερη διάκριση το τομέα από τη εκπαίδευση. αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θέσουμε στόχους. Άρα λέω ότι ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να δοθεί 10% της επίσημης ψυχικής βοήθειας για την εκπαίδευση μέχρι το 2024 και 15% μέχρι το 2030. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό. Να ζητήσουμε δηλαδή από την Κομισιόν να, να επικαιροποιήσει την ανακοίνωσή της επίσης το 2002, την ανακοίνωση για την εκπαίδευση. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα θα απαιτηθούν νέες καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης ε, πέραν της κρατικής βοήθειας, της επίσης ανταξιακής βοήθειας και εκεί πρέπει να τοποθετηθούμε, αλλά να δείξουμε και μεγάλη σύνεση. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την αυτή χρηματοδότηση και ιδίως ε, σε σχέση με ορισμένες πρωτοβουλίες. Κάποιες φορές μπορεί να είναι ανταγωνιστικές με τα ίδια ισχύοντα. Πρώτο, με αναπτυξιακή βοήθεια. αιρεότητα της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να είναι οι στόχοι επίσης πρέπει να καθοριστούν, αλλά και η ε, γραμμή, αν θέλετε, της Κομισιόν. Επίσης, προτεραιότητες. Γιατί υπάρχει ένα χάος σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες. Μίλησα με τον Αρμόδιο Επίτροπο. Το θέμα της απασχολησιμότητας και της βασικής εκπαίδευσης, στοιχειώδους εκπαίδευσης. Εγώ είμαι υπέρ της απασχολησιμότητας και, την, και υπέρ της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχει ο ιδιωτικό τομέα. Άρα δεν υπάρχουν ε, ιδεολογικέ ε, διαφορέ που να μα χωρίζουν. Ε, μιλάμε για μια καθολική εκπαίδευση για όλου, η οποία πρέπει να είναι δωρεάν. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και ιδιωτικά εκπαιδευτικά στήματα. Υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία σε όλε τι χώρε και οι γονεί πρέπει να έχουν την επιλογή. Δεν μιλάμε για μονοπόλιο. Όμω το δικαίωμα στην παιδεία, όπω αναφέρεται και στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ε, επιβάλλει να είναι η εκπαίδευση δωρεάν, να είναι μια καθολική, μια οικομενική υπηρεσία, γιατί είναι μια βασική. Μιλάμε για τη βασική εκπαίδευση. Έχουμε θέσει δύο προτεραιότητες, αρκετά παραδοσιακές. Δεν σε βάστες πάντα όμω. Πρώτον, βασική εκπαίδευση που θα είναι ποιοτική και για όλους. Δεν θα πρέπει κανεί να αποκλείεται ούτε τα κορίτσια, ούτε τα άτομα με αναπηρία και δεν πρέπει να υπάρχουν άλλου είδου διακρίσει, εθνοτικέ, φιλετικέ κτλ. Και δεύτερη ε, προτεραιότητα, ενισχυμένη στήριξη στι χώρε ε, που είναι λιγότερο προηγμένε. Νομίζω ότι αυτέ είναι οι δύο μείζονε προτεραιότητε που πρέπει να έχουμε. Βασική εκπαίδευση, γιατί αν δεν υπάρχει ένα κατόφλι, ε, ένα βάθρο, δεν μπορεί να χτίσει πάνω σε τίποτα από εκεί πέρα. Το είπε και η πρόεδρός μας επίσης, ότι σε κάποιες χώρες Πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει αν δεν έχει τις βασικές γνώσεις, δεν γράφει, δεν διαβάζει. Επομένως η βάση είναι το πάνω, τα θεμέλια. Και έπειτα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι λιγότερο προηγμένες χώρες, ποιες είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη της βοήθειας αυτής. Και βέβαια θα πρέπει εδώ πολύ ξεκάθαρα να πούμε, και το κάνω στην έκθεσή μου, όλοι συμφώνησαν μέχρι τώρα, στο ότι το ίμιση τη βοήθεια για την εκπαίδευση πρέπει να πάει για τη βασική, τη στοιχειώδη εκπαίδευση. 40% τη βοήθεια τη Ένωση προ τι λιγότερο προηγμένε χώρε, ανεπτυγμένε χώρε. Νομίζω ότι αυτό είναι ο δεύτερο ε, άξονα. ερώτα στην εκπαίδευση, στη βασική εκπαίδευση. Ε, πρέπει όμω να έχουμε κάποιε βασικέ γραμμέ για να μην διαχυθούμε ε, ούτε να υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεταξύ των στόχων, ούτε ε, και να είμαστε μεθοδικοί. Έπειτα, ποιότητα της βοήθειας θα πρέπει να αναπτύξουμε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ένα σύστημα αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τη ουσία. Είχε μπει σε δεύτερο πλάνο ε, και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ούτε να έχουμε αποτελέσματα ε, εκπαιδευτικά. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πολύ καλύτερα τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η έρευνα, η ομαδοποίηση δεδομένων, τα, τα εργαλεία αξιόλως πρέπει να είναι όλα αυτά αξιόπιστα. Επίσης, και όλοι οι συνομιλητές μας ε, πρόγραμμα για την εκπαίδευση κομισιών, Παγκόσμια Τράπεζα ε, και Εθνική αναπτυξη και Φορείς μας το είπαν, πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός παρότι βελτιώνεται ήδη των χρηματοδοτών στο πλαίσιο τοπικών ομάδων. Τέλος, αυτό προτείνουμε εμείς και θα υπάρξει συζήτηση. Οι ενώσεις έχουν καταθέσει τροπολογίες σε ορισμένους συναδέλφους, τους έχουν ε, δώσει. Θέλουμε να υπάρχει δημοσιονομική υποστήριξη. Εγώ είμαι υπέρ τη δημοσιονομική υποστήριξη. Δεν μπορούμε ε, να αφήσουμε στι ανθρωπιστικέ οργανώσει. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη να έχουν ένα σύστημα εκπαιδευτικό. Αλλιώ δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα, δημοσιονομική υποστήριξη. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Αλλά φυσικά υπό προποθέσει. Είπα, αξιολόγηση, διαφάνεια, συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και με κάποιες βασικές γραμμές και κάποιες βασικές προτεραιότητες, εκπαίδευση των εκπαιδευτών κτλ. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δημοσιονομική στήριξη λοιπόν ο και αφετέρου όταν, ε, όταν γίνεται βέβαια δημοσιονομική στήριξη και από την άλλη το βλέπουμε τι διαφορά υπάρχει με την υγεία. Πρέπει και εδώ να ευνοήσουμε την εταιρική σχέση παγκοσμίω για την εκπαίδευση. Και αυτό διότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναπτύξουμε τους πολυμερείς οργανισμούς οι οποίοι όλο και καλύτερα λειτουργούν σήμερα. Συνεπώς, αυτή την βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας υπάρχει αναγκαιότητα καλύτερης αξιολόγησης, δημοσιονομικής στήριξης και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολυμερών οργανισμών που πιστεύω ότι πρέπει να θεωρηθούν η προτεραιότητα. Αυτό όσον αφορά τους βασικούς άξονες της έκθεσης. Συνεπώς θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχετικά ομόφωνο μήνυμα, έτσι δεν είναι ιδεολογικό το θέμα νομίζω, αλλά και ένα απλό μήνυμα. Θέλουμε η εκπαίδευση να αποτελέσει προτεραιότητα. Στην εκπαίδευση πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε κυρίως την βασική εκπαίδευση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και άρα πρέπει να βελτιώσουμε όχι μόνο τα ποσά αλλά και την ποιότητα της αρρωγής με δημοσιονομική στήριξη και με την δέσμευσή μας υπέρ της πολυμερούς χρηματοδότησης. Νομίζω ότι ήδη έτσι έχουμε αρκετά στοιχεία. Από εκεί και πέρα και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε φυσικά και για την έκτακτη βοήθεια, για τις ειδικέ ανάγκες, για την υγεία. Εννοείται πρέπει, για να μας κατηγορήσει κανείς, να καλύψουμε όλα τα πεδία. Αλλά να είμαστε επικεντρωμένοι. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους ε, οι οποίοι εμπλούτησαν το κείμενο. Μέχρι το στάδιο των τροπολογιών τέλη Αυγούστου θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα και το φθινόπωρο το Κοινοβούλιο έτσι να μπορέσει να ψηφίσει μια έκθεση που να μπορεί να είναι και χρήσιμη αλλά και δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην ε, θητεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν υπάρχουν πολλέ τροπολογίε. Είναι εύκολο κανεί να κάνει τροπολογίε σε ένα τέτοιο κείμενο, γιατί ψηφίζει κάποιοι, προσθέτει κάποιε λέξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί το κείμενό μα. Αν έχουμε υπερβολικά πολλέ τροπολογίε, δεν περνάει ένα σαφέ μήνυμα. Αντίθετα, κάπω ε, αμβλύνεται το μήνυμά μα, χάνει την ουσία του. Υπάρχουν ε, σήμερα ιστοσελίδες που ζητούν, ε, μάλλον που καταγράφουν τον αριθμό των τροπολογιών ε, που έχουν υποβάλει οι βουλευτές σε κάθε έκθεση. Λες και αυτό, από αυτό εξαρτάται το συμπέρασμα για το πόσο καλά έχουν δουλέψει. Όμως το κείμενο καταλήγει να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έγινε αυτό στις γυναίκες εκεί. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε τα πάντα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 Είπατε ότι θέλετε να υπάρξει ή δυνατόν ομοφωνία ή πλειοψηφία. Δεν θέλουμε όμως ε, να... Ε, θέλω να πω, έχω την εμπειρία ότι αν περιοριστούμε σε κάποια βασικά μάντρα και σλόγγαν υπάρχει ε, μεγάλη πιθανότητα φυσικά να υπάρξει ομοφωνία ή πλειοψηφία υπέρ αλλά μετά τι γίνεται με τις λεπτομέρειες και υπάρχουν κάποιες ε, επαναλήψεις ε, που ε, αν επαναληφθούν δεν νομίζω ότι αυτό είναι θετικό αυτά τα οποία πρέπει να τονιστούν η ε, ε, σχολική, η βασική εκπαίδευση και τα δίδακτρα. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προτεραιότητα για τη δική μου την ομάδα. Η ε, εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά, εκατομμύρια παιδιά που δεν μπορούν ούτε να διαβάσουν ούτε να γράψουν. Η βασική εκπαίδευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό και ε, σε ό,τι αφορά την ε, ε, δημοσιονομική προστήριξη νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε μέσα που θα μπορούν να ορίζουν πολύ ξεκάθαρα την αναπτυξιακή βοήθεια και η ευελιξία δεν πρέπει να είναι ότι ε, θα πρέπει το κράτος ε, που θα παίρνει αυτή τη βοήθεια να την διαθέτει εκεί που θέλει. Απλά τα κράτη που έχουν ε, υποσχεθεί κάτι, να, άμα δεν το κάνουν, να μην παίρνουν αυτά τα χρήματα. και εμείς να είμαστε αυτοί που κάνουμε την ανακατανομή, όχι τα κράτη που λαμβάνουν τα κονδύλα να κάνουν την ανακατανομή. σε ό,τι αφορά την ε, ε, εκ, απασχόληση. Υπάρχουν προβλήματα σε αναπτυγμένες ε, χώρες ε, σε ό,τι αφορά την ε, εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση συγκεκριμένα. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ χειρότερο στις ε, μη αναπτυγμένες χώρες η απασχολησιμότητα, η απόκτηση δεξιοτήτων είναι σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση δεξιοτήτων, πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση και κατάρτιση για να μπορεί πιο εύκολα επιτά κάποιος να βρει δουλειά. Επίσης πρέπει να είναι ποιοτική και για όλους η εκπαίδευση εκπαίδευση. Αλλά να μην χάσει και τη σημασία του αυτό. Σε ό,τι αφορά το διοικητικό κλάδο, ότι πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική πλευρά. θα πρέπει να μπορεί ε, να υπάρχει μια ε, να πρέπει να υπάρχει απόκτηση διοικητικών δυνατοτήτων, αλλά να υπάρχει ένα αντιστάθμιζα, να ε, μπαίνει αυτή η βοήθεια ε, σε πρακτική μετά. Να μην χρειάζεται για 50 χρόνια να συνεχίζει να παρέχεται διοικητική υποστήριξη για την οργάνωση της διοικητικής δομής κυβέρνησης. Θα πρέπει η εκπαίδευση να στοχεύει στο να μπορεί οι ίδιοι ε, να αναπτύξουν τις δικές τους δομές ώστε να μην υπάρχει και φυγή εγκεφάλων έπειτα. Νέες τεχνολογίες, ε, επίσης είναι σημαντικό, το είπε ε, και οι εισηγητές, πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση. Είχαμε πει πρόσφατα ένας υπολογιστή αναπαιδεί. αλλά ε, πρέπει να πω ότι υπάρχουν νέες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν είναι καθόλου θέμα ιδεολογίας. Η αριθμητική δεν ε, ε έχει να κάνει με ιδεολογίες. Με ιδεολογίες ε, είναι πρακτικά πράγματα. Ε, τα πράγματα είναι πολύ απλά σε όλες τις χώρες. Ε, ο πίνακας και η κοιμωλία ε, υπάρχουν παντού. Και επίσης η εκπαίδευση στον τομέα της υγείας επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ενισχύσουμε τις δεξιότητες, να υπάρχει πληροφόρηση στον τομέα της υγείας, πρέπει να υπάρξει μια, ένας πολλαπλασιασμός των θέσεων εργασίας και να μπορούν οι εργαζόμενοι να αποκτούν νέες δεξιότητες, οι οποίες θα εκμεταλλευτούν. Και εκπαιδευτικές μέθοδοι ε, και ε, το One Laptop Per Child και αυτό που δεν ανέφερε το επιπρόεδρος όμως ε, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δώσουμε επίσης ε, έμφαση στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς ε, και η αξιολόγηση, το είπε και πρέπει να αξιολογούμε και τα συστήματα τα αλλά και τις επιδόσεις. Δεν πρέπει να προχωρούν αυτοί οι οποίοι έχουν γονείς που μπορούν να δωροδοκίσουν κάποιον, αλλά αυτοί που είναι ικανοί και πρέπει να ε, βάλουμε πιστεύω πιο ε, ψηλά τον πύχη για τις χώρες αυτές. Και ένα τελευταίο, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ε, είναι όλοι πολύ σημαντικοί. Αλλά βλέπουμε ότι σε κάποια ε, κράτη υπάρχουν δυσκολίες με κάποιους συγκεκριμένους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι για τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε κάποιες χώρες. Θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε και πού πρέπει να δώσουμε το βάρος. Θέλουμε δηλαδή να προωθήσουμε όλους τους στόχους ή να κάνουμε κάποια επιλογή. Επίσης ε, πρέπει να υπάρξει ε, σεβασμό σε όλες τις θρησκείες, ε, να, υπάρξει, να μην υπάρχει καμία διάκριση για λόγους φύλου, εθνότητας κτλ. Το θέμα είναι όμως η ίδια η κοινωνία σε κάθε χώρα που μπορεί να εστιάσει πώς μπορεί να υπάρξει μια χειραφέτηση για θέματα που εμάς μας φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και κύριε Χαουτάλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ και για την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα στις συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών πριν καταλήξουμε στην υποβολή τροπολογιών. Ήταν πολύ σημαντικό και όπως ε, είπατε, ίσως θα πρέπει να πειραματιζόμαστε πιο συχνά με αυτή τη μεθοδολογία. Τώρα, αυτά που εκτιμώ όλου ιδιαίτερω στο σχέδιο έκθεση είναι τα εξή. Δίνουμε προτεραιότητα στη βασική ε, εκπαίδευση στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε που σημαίνει 40% της εκπαιδευτικής αρρωγής τώρα. Δημοτικό και γυμνάσιο θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλους. Πολύ καλά αναφέρεται και αυτό στην έκθεση. Και χαιρόμαστε που γίνεται και έκκληση στις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην στηρίξουν την ιδιωτική εκπαίδευση. Τουλάχιστον να μην υπάρχει δημόσια στήριξη σε αυτήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφέρετε επίσης τη διαρροή εγκεφάλων και την δυνατότητα ε, να προωθήσουμε την ε, κυκλική κινητικότητα. Εννοείται ότι δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε με την τεχνολογία τους δασκάλους, έτσι, κάτι που γίνεται μερικές φορές. Και επίση πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ζητήσουμε αύξηση τη συμμετοχής στην παγκόσμια εταιρική σχέση για την εκπαίδευση εκπαίδευση. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η παγκόσμια εταιρική σχέση για την εκπαίδευση φαίνεται να είναι μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα επιτυχής. Καταφέρνει να οικοδομούνται πραγματικά εκπαιδευτικά συστήματα. Δεν πρόκειται απλώς δηλαδή για την οικοδόμηση κτηρίων, σχολείων. Όχι. Έχει να κάνει και με τις ε, πραγματικές ανάγκες του συστήματος. Ο κύριο Βίλαν πολύ σωστά είπε ότι και η κατάρτιση των διδασκόντων είναι στοιχείο κλειδί. Γιατί στη χώρα μου τουλάχιστον η ποιότητα της εκπαίδευσης οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ε, καταρτούνται ικανοποιητικά οι εκπαιδευτικοί και χαίρουν μεγάλης εκτίμηση στην κοινωνία. Έχει αλλάξει αυτό. Δεν ήταν έτσι παλιά. Κάτι το οποίο επίσης είναι βασικό για να πετύχουμε αλλαγές είναι και το θέμα της εκπαίδευσης σε θέματα σεξουαλικότητας. Πρέπει να αναφερθεί και αυτό πιστεύω. Λοιπόν, εντάξει, υπόσχομαι, δεν θα υπάρχουν πολλές τροπολογίες, αλλά δύο-τρεις θα τις υποβάλω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να σχολιάσει, να είστε το... Α, εσείς, παρακαλώ, η νέα μας ε, αντιπρόεδρος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω φιλανδικά, τη μητρική μου γλώσσα, αν μου επιτρέπετε. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ με αυτά που ακούστηκαν. Εγώ είμαι δασκάλα το επάγγελμα Τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια δούλεψα ως δασκάλα στη Φινλανδία με παιδιά της, ε, του Δημοτικού και πιστεύω ότι η εκπαίδευση αλλά και η επαγγελματική κατάρτιση έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η προαγωγή της εκπαίδευσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντική και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η τεχνολογία αλλά πάλι ε, όταν γίνονται πρόοδοι δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν πάντα οι τελευταίες ε, ε, τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα διαθέσιμα. Προχωρούμε όμως παρόλα αυτά. Είναι μεγάλη, πρόοδος, η μεγάλη πρόκληση λοιπόν, να το πιστεύω, 10% των ε, δημοσίων κονδυλίων ε, μέχρι το 24 και 15 έως το 30 για την εκπαίδευση είναι μια μεγάλη πρόκληση. Μακάρι να υλοποιηθεί, θα χαρώ πολύ. Ε, αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικά τα, σημαντικό να υπάρχουν ρεαλιστικά εθνικά προγράμματα. Δεν μπορούμε να εξαγάγουμε την ε, πολιτική, την εκπαιδευτική που έχει μία χώρα σε άλλες χώρες και τις ε, χώρες της ανάπτυξης. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να βρούμε τρόπους για διαμόρφωση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων με βάση τις δυνατότητες που έχει κάθε χώρα. Πάντα γίνεται βέβαια λόγος για ε, εκπαίδευση ανοιχτή σε όλους, που δεν θα αποκλείει κανέναν. Τα γόρια και τα κορίτσια δηλαδή πρέπει να στηριχθούν, να στηριχθούν εξίσου, να στηριχθούν και οι μειονότητες, ε, να μην λησμονηθούν τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και δι με πνευματική αναπηρία. Και βεβαίω η επιμόρφωση των διδασκόντων, αναφέρθηκε και νωρίτερα, στη Φινλανδία, στο φινλανδικό πρότυπο, έχει τεράστια σημασία. Ε, έχουν ε, πανεπιστημιακό δίπλωμα η εκπαιδευτική, πράγμα το οποίο μπορεί να μην ισχύει σε κάθε χώρα, αλλά γενικά το προσωπικό στον χώρο της εκπαίδευσης χρειάζεται και την ε, εκπαίδευση κατάρτιση και την επιμόρφωση. Είναι κάτι λοιπόν το πολύ σημαντικό η επιμόρφωση και όπως είπα με ιδιαίτερη έμφαση στους δασκάλους και η επαγγελματική κατάρτιση. Βέβαια εδώ ε, πρέπει όταν συζητούμε τα θέματα αυτά να μην μιλούμε μόνο για τον τομέα τον ιδιωτικό. Πρέπει να μιλούμε και σε επίπεδο αναγκών και προοπτικών για τον δημόσιο τομέα, για την κρατική εκπαίδευση. Ε, μην λησμονούμε τι είδου ανάγκες θα έχουμε σε επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ε, και θέσεις εργασίας. Η Φινλανδία, παραδείγματι, θα έχει ανάγκη σε εργατικό δυναμικό ε, για τον τομέα τη της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και άλλους τέτοιους τομείς του δημόσιου τομέα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε ρητά να αναφερθούμε στο θέμα της ε, υγείας. Την ανάγκη να προσφέρεται η ε, προληπτική ιατρική φροντίδα στο σχολείο για όλα τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μια βασική πρόνοια ιατρική που μπορεί να προσφέρεται κάποιες βασικές εξετάσεις ιατρικές θέματα των εμβολιασμών μπορεί να παρακολουθούνται μέσα από το σχολείο, να προσφέρονται τα εμβόλια στο σχολείο. Αυτά, ευχαριστώ. Αυτά θα θέλω να μπουν στην έκθεση. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Δεν ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Ε, θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω το θέμα των ε, μη καθαρών, το μη, ε, το εφανών εξόδων, γιατί πολλές φορές έχω επισκεφθεί περιοχές και σχολεία που είναι υποτίθεται, όπου είναι υποτίθεται δημόσια η εκπαίδευση. αλλά πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κρυφά έξοδα αυτό οφείλεται ακόμα και στο γεγονός ότι είναι πολύ χαμηλή η αμοιβή των διδασκάλων παραδείγματι και άρα χρειάζεται κάποια υποστήριξη ή σε, άλλους, ε, ε, σε άλλες χώρες όπως είδαμε στην Ουγγάντα στην αποστολή μας με το να υπάρχει υποχρεωτική στολή σχολική ε, επιβαρύνονταν η οικογένειά τους με ένα σημαντικό έξοδο. Άλλο που είδαμε σε αποστολή που ακούστηκε νωρίτερα ότι έχει τελειώσει η εποχή του πίνακα και της κοιμωλίας. Δεν υπήρχε καν σχολικό κτίριο. Το σχολείο των παιδιών ήταν ένα, ε, δέντρο. Και γύρω από το δέντρο αυτό τα παιδιά έκαναν ε, το μάθημά τους. Ή άλλο παράδειγμα που επισκέφθηκα ένα σχολείο με 150 παιδιά στην τάξη και μιλούσα με τον δάσκαλο και του ζήτησα ένα μολύβι για να γράψω κάτι, ένα στυλό και μου δάνει το στυλό του και μετά εγώ αφηρημένη όπω θεώρησα ότι ίσως είναι το δικό μου, ούτε καν σκέφτηκα, πήγα να το βάλω στην τσάντα μου και είδα τον τρόμο στα μάτια του δασκάλου γιατί δεν είχε άλλο στυλό να γράψει και χρειάστηκε να μου θυμίσει να του δώσω το στυλό του. Στην Κένια σε μια παραγκούπολη με εξαιρετικό δάσκαλο, εξαιρετικούς δασκάλους, γιατί θα συμφωνήσω εδώ η ποιότητα των διδασκάλων σε τόσο σκληρές συνθήκες και όταν βλέπουμε στο αποτέλεσμα που έχουν στα παιδιά με το, με το πολύ καλό του εκπαιδευτικό επίπεδο κτλ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να του προσφέρουν, αλλά βέβαια όσο πιο μακριά είμαστε από τα κέντρα των πόλεων, τόσο πιο δύσκολε είναι οι συνθήκε στην επαρχία, στην ύπεθρο κτλ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και χαίρομαι που μπορούμε να τα συζητήσουμε πριν να κλείσει η θητεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα. Ρένε Μαλή, DG DEFCO, Judith Μπάρνα από την ECO. Ας ακούσουμε πρώτα την DEFCO και μετά την ΕΚΟ. Χρηματοδότηση μειούμενη για την ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τι νέα εργαλεία έχετε υπόψη, θα ήθελα να μας πείτε. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Χαίρομαι που ακόμα και στα μέσα Ιουλίου έχουμε τόσους πολλούς ε, ε, παρόντας εδώ στη συνεδρίαση. Ρενέ Μάλι είναι το όνομά μου. Στην ΤΕΦΚΟ ασχολούμαι με τα θέματα της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχω και τη συνάδελφο από την ΕΚΟ αλλά και τη συνάδελφο από την ε, ομάδα μου εδώ στα δεξιά μου και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή έκθεση που έρχεται και την κατάλληλη στιγμή. Ε, ιδιαίτερα εκτιμούμε την ανάλυση, ιδιαίτερα θετικά εκτιμούμε την ανάλυση και την έμφαση που δίδεται στην προαγωγή της εκπαίδευσης για τους σκοπούς της, της ανάπτυξης. Πιστεύουμε όντως ότι είναι ο ευφιέστερος τρόπος αναπτύξεως. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και για κάθε άλλο ε, στόχο αναπτυξιακό ε, έχει τεράστια σημασία 640 εκατομμύρια παιδιά δεν πάνε σχολείο. Πολλά από τα, σχολεία, τα παιδιά που πάνε σχολείο δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση. Ευχαριστούμε για τις, για τις εικόνες που μας μεταφέρατε με τα παιδιά που κάνουν μάθημα γύρω από ένα δέντρο. Επομένως, ε, είναι πολύ σημαντικό το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ασχολείται με το θέμα αυτό την εκπαίδευση και οπωσδήποτε πρέπει να χορηγηθούν και περισσότερα εργαλεία, πρέπει να επικαιροποιηθεί η σχετική πολιτική. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση αυτή της έκθεσης. Επίσης θεωρούμε ότι η έμφαση στην πρωτοβάθμια, αλλά και στις, ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, έχει στη σημασία. Άλλωστε αυτό κάνουμε και εμείς στη δουλειά μας. Άλλωστε κάνουμε και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων με το που ξεκινάμε τη συνεργασία με τις ε, χώρες εταίρους. Θα ήθελα παρεπιπτόντως να επισημάνω ότι και στην πολυμερή βοήθεια την παγκόσμια συνεργασία δηλαδή για την ε, εκπαίδευση αλλά και στις ε, διμερείς σχέσεις μας πάντοτε στρεφόμαστε και εξετάζουμε με τρόπο συστημικό το σύστημα, το εκπαιδευτικό, να είναι και ισότιμη η πρόσβαση και ποιοτική η εκπαίδευση που προσφέρεται. Και ευχαριστώ πολύ για την ενθάρρυνση που μας δώσατε να συνεχίσουμε τις επαφές. Αυτό, όπως είπα, γίνεται και στις πολυμερείς και στις διμερείς, αλλά και σε σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα, με τους, ε, συνεταίρους, με τους εταίρους σε, σε πολυμερές επίπεδο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είμαστε και οι μεγαλύτεροι εταίροι σε όγκο προσφερόμενης βοήθειας. Επομένως και έχει πει ο Επίτροπο ότι θα συνεχιστεί η στήριξη της παγκόσμια εταιρική σχέσης για την εκπαίδευση και στην ε, επόμενη, στον επόμενο δημοσιονομικό σχεδιασμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, ένα πολύ σημαντικό για μας επίσης σχόλιο ήταν ε, η ενίσχυση της, του δυναμικού απορρόφησης, αυτό που αναφέρθηκε και από εσά σε ορισμένες χώρες εταίρου, έχει κρίσιμη σημασία. Έχει να κάνει βέβαια με τι διατυπώσεις τη υλοποίηση. Θέλουμε να προσφέρουμε τη βοήθεια όταν είναι δυνατόν να απορροφηθεί, να γίνει αποδεκτή, όταν υπάρχουν κατάλληλε συνθήκες ή προχωρεί προ τι κατάλληλε συνθήκε η χώρα εταίρο. Ε, εκείνες που θα του επιτρέψουν μια με συγχωρείτε λέει ο, ο μιλητής για το τηλέφωνο. Ε, όταν θα έχει προχωρήσει προς τις ε, συνθήκες πλαισίου η εν λόγω χώρα και το πλαίσιο για τις δεξιότητες. Πάντοτε οι συνάδελφοι ε, παρακολουθούν και επικαιροποιούν τα πρότυπα για την εκπαίδευση και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν. Η ψηφιοποίηση επίσης μας απασχολεί, την προάγουμε με μεγάλη προσοχή Επίσης ε, η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είτε είναι διμερής είτε είναι πολυμερή τα προγράμματα έχει τεράστια ποσά, 5,5 δις. Και επιπλέον την ε, χρηματοδότηση από την ανθρωπιστική εκπαίδευση μέσω της ΕΚΟ που πάει σε διμερή, ανώτερη και πολυμερή, ε, εκπαίδευση και πολυμερή προγράμματα. Στην έκθεση θα θέλαμε ίσως να δούμε και ίσως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί αρκετά σαφώς εν μέρει αναφέρθηκε αυτό το η στόχη της ε, ανάπτυξης 4,7 και ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση είναι κάτι που συζητούμε και με τις ε, κυβερνήσεις με τις οποίες έχουμε εταιρικέ σχέσεις. Κοιτούμε τα προγράμματα σπουδών, κοιτάμε να δούμε αν προάγουν ή όχι τα, τα προγράμματα αυτά σπουδών, τις ιδέες της ε, ε, διαλλακτικότητας, της διαφοράς, της ανοχής του άλλου. Η διάσκεψη αναφέρθηκε, η ενίσχυση της ισότιμης εκπροσώπησης στα σχολεία, αναφέρθηκε. Κάτι ακόμη που βλέπουμε είναι μια πολύ περιορισμένη ακόμη απόδοση της ε, επένδυσης εντός εισαγωγικών, γιατί δεν εννοώ οικονομική επένδυση, αλλά κοινωνική απόδοση της εκπαίδευσης για τα ε, μικρά παιδιά. Ε, χρειάζεται λοιπόν περισσότερη χρηματοδότηση, ναι. Χρειάζεται μια κατάλληλη πολιτική, ναι. Χρειάζεται να ενισχυθούν τα συστήματα των χωρών εταίρων μας. Στη χρηματοδότηση υπό το νέο πολιτές νοσονομικό πλαίσιο, ο Επίτροπος το έχει αναφέρει. Και στο παρελθόν 20% του νέων μέσων που προτείνονται θα είναι αφιερωμένα στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Αυτή είναι η βασική ιδέα και πρόταση. Ανάπτυξη του ανθρώπου σημαίνει βέβαια οπωσδήποτε και εκπαίδευση και κατάρτιση. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο Επίτροπος πόσο μεγάλη σημασία έχει η εκπαίδευση και η κατάρτιση και για τους στόχους της ανάπτυξης και έτσι θα συνεχίσει να διαδραματίζει αυτή η εκπαίδευση πολύ σημαντικό ρόλο και στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά είχα εγώ να πω. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να προσθέσουν κάτι σε όρους ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι θα σας αναφέρω κι εγώ κάποια σημεία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή για την στάση του απέναντι στην ε, νέα ανακοίνωσή μας για την προστασία σε περίπτωση κρίσεων. Είπατε ότι δεν είχαμε νέα ανακοίνωση για την εκπαίδευση. Αυτή η ανακοίνωση ίσως να καλύπτει σε ένα βαθμό το κενό. Ίσως βέβαια όχι με το πεδίο εφαρμογή που όλοι θα επιθυμούσαμε. Οπότε για την ανθρωπιστική βοήθεια έχουμε φροντίσει να αυξήσουμε την χρηματοδότηση για να στηρίξουμε την εκπαίδευση και πρέπει να προσέξουμε ότι τα παιδιά κάτω από όλες τις συνθήκες, ακόμα και αυτά τα παιδιά που ζουν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, πρέπει να χαίρουν το δικαίωμα αυτό στην εκπαίδευση. Οι κυβερνήσεις βέβαια ε, μπορεί να μην τα καταφέρουν παρά την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε εμείς να ε, περιλαμβάνουν στην εκπαίδευση όλα τα παιδιά. Άρα αυτό πρέπει να είναι μια προσπάθεια. Και το άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, όπως είπατε κι εσείς, δεν φτάνει. Η ανθρωπιστική βοήθεια, η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι και γι' αυτό και έχουμε και την ανακοίνωσή μας για την προσέγγιση Nexus. Παρά την προσέγγιση της ανακοίνωσης, ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό. Όταν βοηθούμε με ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν παράλληλα κανάλια. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ όλων των προσπαθειών και ο απότερος στόχος μας να είναι η πρόσβαση σε όλα τα παιδιά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Πεγιό, σχόλια. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την ποιότητα των παρεμβάσεών σας σήμερα που μας επιτρέπουν να δούμε ότι ο στόχος είναι κοινό για όλους μας, όπως επίσης και οι προτεραιότητές μας. Θέλω να απαντήσω τώρα σε δύο-τρία προβλήματα τα οποία τέθηκαν από τον ε, Αντιπρόεδρο Βίλαντ, ε, τον Αντιπρόεδρο Χαουτάλα και άλλους συναδέρφους. Το θέμα της τεχνολογίας. Νομίζω ότι εδώ κάνουμε μια λάθος συζήτηση για την τεχνολογία. Εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες όσο μπορούμε και για την κατάρτιση των διδασκόντων, των εκπαιδευτικών. Αλλά η χρήση των νέων τεχνολογιών σημαίνει ότι είναι εκεί για να προσφέρει στήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ή εκπαιδευτικούς θα έχουμε ή νέες τεχνολογίες, όχι, και τα δύο μαζί. Έχουν ήδη γίνει αξιολογήσεις και εννοείται ότι κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούν να προωθήσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, αλλά κοιτάξτε, και εμείς στην ε, Γαλλία προσπαθούμε να αντιγράψουμε το μοντέλο της Φιλανδίας και το πρώτο είναι όντως η κατάρτιση, η επιμόρφωση των ε, διδασκόντων στις νέες τεχνολογίες. Γιατί ένας πειρασμός που υπάρχει συχνά στην Αφρική είναι επειδή ακριβώς ε, δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς να βάζουν τεχνολογία να τους αντικαθιστά. Όχι. Κάτι άλλο σοβαρό και χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Φίλαντ να το λέει. Συμφωνούμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια για την εκπαίδευση έχει ως προορισμό να εκπαιδεύσει τους πολίτες οι οποίοι θα δουλέψουν στη συνέχεια στη συγκεκριμένη χώρα. Και το ζήτημα που τίθεται βέβαια είναι η διαρροή κεφάλων. Επ' αυτού θα λέγω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν πολιτικές ανοιχτές ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται στην Ευρώπη για ένα διάστημα αλλά μετά να επιστρέφουν. Γιατί αν κοπεί αυτό ο διάβλος, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα έρθουν μόνιμα να εγκατασταθούν εδώ. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι κλειστή και έτσι απαντάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ συμφωνώ για αυτό που είπατε με τα πανεπιστήμια και στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να δίνουμε μαθήματα σε άλλες χώρες, όπως κάνουμε, ενώ δεν τους δίνουμε καν τα στοιχειώδη, και μετά να ακούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες αυτά που λένε για την ε, ανοχή, για τη συμμετοχή κλπ. Συμφωνώ μαζί σας. Το πρότεινα στη Γαλλία, δεν έγινε. Λοιπόν, δεν ε, να λέμε να δεχόμαστε στα πανεπιστήμια, Βεβαίω. Και συμφωνώ επίση, και μάλιστα με εκπλήσει που το ξέχασα πριν, την εκπαίδευση για τα μικρά παιδιά. Όσο γίνεται πιο νωρίς, όλες οι μελέτες και νευροψυχολογίας που γίνονται για τη γλώσσα, για την ανάπτυξη κτλ. λένε ότι όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η εκπαίδευση, αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά Πόσο μάλλον για τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα προβληματικά. Οπότε, ναι, και για την ατομική ανάπτυξη και γενικότερα η εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία έχει πάντα θετικά αποτελέσματα. Παντού. Τώρα, κυρία Φατάλα, έθεσε ένα θέμα που όντω δεν πρέπει να το κρύβουμε, το έχουμε συζητήσει με τους άλλους, αλλά πρέπει να το πούμε και εδώ. Το θέμα της δωρεάν εκπαίδευση. Και επανέρχομαι σε αυτό. Κανείς δεν ζητάει το μονοπόλιο. Εννοείται. Είναι πράγματα που συζητήσαμε στην Ευρώπη το 19ο αιώνα. Φυσικά και υπάρχουν ε, και συστήματα ιδιωτική εκπαίδευση παράλληλα με τα συστήματα δημόσια εκπαίδευση. Αν οι γονεί το προτιμάνε, έχει καλώ. Όμως την εκπαίδευση πρέπει να την προσφέρει το δημόσιο, το κράτος, δωρεάν ακριβώς για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν. Υπάρχουν επιχειρήσεις αγγλικές, γαλλικές ε, και άλλες όμως έτσι και από την Ασία που προσπαθούν να αναπτύξουν αυτό το εμπόριο της εκπαίδευσης. Και όχι της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έτσι, πανεπιστημιακής ή ε, όχι, της βασικής εκπαίδευση, της πρωτοβάθμιας. Και είναι σκανδαλώδε. Δεν είναι δυνατόν για να πάνε στο δημοτικό τα παιδιά να πρέπει να πληρώνουν οι γονείς τους. Αυτό ισχύει όμως στην Αφρική. Το θέμα μου δεν είναι ιδεολογικό. Δεν είναι ότι θέλω να κυνηγήσω τον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική εκπαίδευση. Όχι, απλώ λέω ότι η βασική εκπαίδευση θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλες τις χώρες. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μα τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό εδώ από το θέμα της υγείας. Γιατί λέμε, όπως... Μάλλον, μια που δεν έχουν λειτουργήσει καλά ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στην εκπαίδευση με την αναπτυξιακή βοήθεια, βλέπουμε ότι τα ποσά που πρέπει να επενδυθούν είναι τεράστια και επειδή αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσκολίε οι χώρε κτλ, υπάρχει ο πειρασμό να ζητάμε από τον ιδιωτικό τομέα να καλύψει αυτή την αδυναμία. Αλλά θα πρέπει σε 10, 20, 30 χρόνια να ξέρουμε τι μας περιμένει αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο ε, που να έχουμε ιδιωτική εκπαίδευση αντί για δημόσια στη βασική εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε στην έκθεση, εξηγώντας ότι δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μπορεί να υπάρχει επιπληρωμή ε, μόνο βασική εκπαίδευση. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ υπερβολικά, χαίρομαι που συμφωνώ με τις προτεραιότητες, όλοι συμφωνούμε, το βλέπουμε. Επίσης και για τη σύνδεση αυτή με την υγεία. Θα βρούμε με ποιο τρόπο να το πούμε σε κάποιες χώρες δεν είναι εύκολο στα σχολεία, οπότε δεν ξέρω πώς θα γίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στα σχολεία να μπορεί να υπάρχει κάποια πρόληψη, αν μη τι άλλο. Θα βρούμε τον τρόπο να το βάλουμε. Και συμφωνούμε, και είναι πολύ βασικό πέρα από τις προτεραιότητες, δηλαδή βασική εκπαίδευση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, συμφωνούμε και για το θέμα της δημοσιονομικής στήριξης μέσω της πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση εταιρικής σχέσης. Αλλά πρέπει να δούμε το θέμα των προϋποθέσεων της αιρεσιμότητας. Δηλαδή, ναι, δημοσιονομική στήριξη, ώστε να φτιάξουν τα συστήματά τους οι χώρες, αλλά προσοχή, τα χρήματα να χρησιμοποιούνται σωστά. Οπότε να βάζουμε προϋποθέσεις για τον τρόπο, για το περιεχόμενο, δεν ξέρω, κάποιες προϋποθέσεις, ε, τα ακούσαμε. Αυτά. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που οργανώσατε την ε, συζήτηση τώρα πριν τις διακοπές και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για την ποιότητα των παρεμβάσεών σας. Θα συνεχίσουμε και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μία έκθεση που θα έχει την πυκνότητα που θέλουμε γιατί αυτό που είπατε εγώ δεν θα ξανάρθω στην επόμενη θητεία, αλλά κάτι βασικό για την Ευρώπη είναι ότι οι εκθέσεις που κάνουμε, που εκπονούμε, δεν πρέπει να γίνονται για αυτό σκοπό, δηλαδή για να ικανοποιούμε εμείς, θα πρέπει αυτοί απ' έξω να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Γιατί στο τέλος θα καταλήγουμε να ψηφίζουμε εκθέσεις που κανένας δεν θα διαβάζει. Γιατί πρέπει να τον αγνωρίσουμε ότι δεν είναι πάντα ευανάγνωστες οι εκθέσεις μας. Γι' αυτό λοιπόν το κείμενο αυτό να το κρατήσουμε έτσι ώστε να προβάλλεται το μήνυμά μας. Και ευχαριστώ την κυρία Χαουτάλα για τις προσπάθειές της. Και αυτό που είπατε για τη σεξουαλική εκπαίδευση, ναι, όντως. Και αυτό θα το λάβουμε υπόψη μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κρίμα που δεν θα ξανάρθετε στην επόμενη θητεία, κύριε Πηγιό. Κάτι τελευταίο. Όταν μιλήσατε για τον ιδιωτικό τομέα, Πρέπει να πάρουμε τα μαθήματά μας από τα όσα έχουν δοκιμαστεί μέχρι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Χτίζονται σχολεία. Υπάρχουν και σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Αλλά μερικές φορές καταλήγετε να πληρώνετε περισσότερα από ό,τι αν είχατε δανειστεί χρήματα. Η χώρα μου, η κυβέρνησή μου το έκανε. Χρησιμοποίησαμε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και τώρα το ξέρω από τα σχολεία στη δικιά μου την πόλη ότι πρέπει να ξεπληρώνουν δάνεια τα οποία τελικά είναι πολύ πιο ακριβά από ότι αν το ίδιο το κράτος είχε χτίσει τα σχολεία αυτά. Οπότε, μετά τι γίνεται, αναγκαζόμαστε να πάμε στις τράπεζες, να διαπραγματευτούμε με τις τράπεζες στις οποίες ανήκουν τα δάνεια. είναι ένα τελικά πολύ ακριβό μοντέλο μακροπρόθεσμα. Φυσικά βραχυπρόθεσμα είναι πολύ ωραίο γιατί ορίστε έχεις ένα καινούριο σχολείο λαμπερό. 10-15 χρόνια μετά όμως το χρέος είναι τόσο μεγάλο και έρχονται άλλοι απ' έξω και ελέγχουν τι κάνεις εσύ στο σχολείο σου. Οπότε ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ το πήρα αυτό το μάθημα. Δεν υπάρχουν βέβαια μαγικές λύσεις, έτσι. αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα. Γίνονται δοκιμές, ας παίρνουμε τα μαθήματά μας. Και μην βάλουμε τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου να κάνουν τα ίδια λάθη που έχουμε κάνει εμείς. Ωραία. 3 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Να μην υπάρχουν πάρα, πολλές τροπολογίες και να τα πείτε και στους άλλους συναδέλφους, παρακαλώ. Ίσως θα πρέπει να είμαστε σκληροί. Μερικέ φορέ αν δεν είμαστε σκληροί θα πρέπει να λέμε όχι, όχι, όχι. Αν θέλετε να κρατήσετε την έκθεσή της με την ουσία της, ε, να πείτε όχι στις τροπολογίες που θεωρείτε. Ξέρω ότι είναι σκληρό, αλλά τέλος πάντων, η Χέντι. Οι συντονιστές θα πρέπει να στηρίξουν αυτή την ιδέα της πρώτης ανταλλαγής πριν η υπάρξη υποβολή τροπολογιών είναι χρήσιμο. Θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε πιο συχνά αυτόν τον μηχανισμό. Ναι, λέει πρόεδρο, πολύ καλή ιδέα. Θα προσπαθήσουμε. Στην επόμενη θητεία θα προσπαθήσουμε. Έχω ήδη προσπαθήσει να αλλάξω τους κανόνες πριν από καιρό. Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα, αλλά πρέπει να φύγω νωρίτερα από ό,τι περίμενα εξαιτία όλων των προβλημάτων των κυκλοφοριακών, τη διάσκεψη στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να φύγω νωρίτερα. Οπότε θα αναθέσω την Προεδρία στη νέα Αντιπρόεδρο. Εύχομαι σε όλους σας καλές καλοκαιρινές διακοπές. Προσωπικό, ευρωβουλευτές, βοηθούς, προσκεκλημένους και στους διερμηνείς βέβαια, λέει η Πρόεδρος, που ξέρω αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες. Ωραία, τέλη Αυγούστου θα τα ξαναπούμε. Και παραδίδω την Προεδρία στη νέα Αντιπρόεδρο. Παρακαλώ. Okay, then. Shall we start? Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. We are opening the agenda number 13. And it's 24th conference of the Περνάμε στο επόμενο σημείο, 24η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Κάθε χρόνο υπάρχει διάσκεψη των μερών της ε, Σύμβασης Πλαισίου των Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Το 2015 το αποτέλεσμα της ε, διάσκεψης αυτής ήταν η σύναψη της Συμφωνίας των Παρισίων. Και τώρα, φέτος, θα πρέπει να συμφωνηθεί ε, οι κανόνες, ένα rule book για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας των Παρισίων. Η 24η διάσκεψη των μέρων, η COP24 δηλαδή, θα γίνει στο Κατοβίτσε, στην Πολωνία. και θα είναι η ε, ευκαιρία για να ε, μελετηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο μέτωπο της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής ε, και ελπίζουμε να ενισχυθεί η σχετική δράση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων έχει συντάξει ένα σχέδιο ψηφίσματος στο πλαίσιο της προπαρασκευασίας προπαρασκευής για την COP24. Θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 10 Οκτωβρίου αυτό το σχέδιο. Συντονιστές Επιτροπής ΔΕΒΕ αποφάσισαν τον Απρίλιο πως η Επιτροπή μας θα συνεισφέρει με γνωμοδότηση αυτό το ψήφισμα, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν γνωμοδοτήσεις, σε προτάσεις ψηφίσματος για τις οποίες δεν υπάρχει έκθεση. Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνατότητα άλλη, ώστε να μπορέσει ε, να συμβάλλει σε, στην κατάρτιση μιας πρώτης ψηφίσματος κάποια άλλη επιτροπή πλήν της καθήλυνα Χθε οι συντονιστές μας αποφάσισαν το εξή. Θα καταθεθεί από την Επιτροπή μας σε μία δέσμη τροπολογιών θα την εγκρίνουμε μετά τις θερινές διακοπές και θα την αποστείλουμε στην Προεδρία της Επιτροπής ΕΝΒΗ για να συμπεριληφθεί στην δική τους ψηφοφορία, στην ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματός τους. Αυτή η διευθέτηση είναι παράλληλη με μια αντίστοιχη διευθέτηση μεταξύ Επιτροπής Ήτρε και Επιτροπής Ένβη. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσουμε την κυρία Μακλίν. Είστε εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Μακλίν και εργάζομαι για το δίκτυο περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών με κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό ότι προσκαλείτε την κοινωνία των πολιτών ε, στην Επιτροπή σας ώστε να συμβάλλουμε στην προετοιμασία της ΔΕΒΕ για το ψήφισμα της ε, ΚΑΠ24, COP24 και στις κλιματικές δράσεις βεβαίως ε, δραστηριοποιούμαστε, αλλά θα μιλήσω σήμερα για τα αναπτυξιακά περισσότερα και τι μπορούμε να περιμένουμε από την COP24 ε, της Πολωνίας φέτος. Τρία χρόνια μετά την έγκριση συμφωνίας των Παρισίων το 2015, Έχουμε νομίζω πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα. Το μεγαλύτερο από αυτά για την επόμενη διετία λίγο πολύ είναι η COP24 της Πολωνίας. Γιατί, γιατί στόχος είναι να συμφωνήσουμε στις ε, κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο οι συμφωνίες, ε, η Συμφωνία των Παρισίων σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο συγκεκριμένα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον λόγο αυτό να έχουμε την ε, ε, τις προτάσεις ε, που θα κατατεθούν από την οπτική σκοπιά της ανάπτυξης για τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, για την προαγωγή των δικαιωμάτων και όλα αυτά και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η συμβολή, η συμμετοχή στη διαδικασία της Επιτροπής σας με τις τροπολογίες που θα καταρτήσει. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε από την ε, ΚΑΠ 24 όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα και από τον ε, Πρόεδρο στόχος είναι να βρεθεί ο τρόπος να υλοποιηθούν οι στόχοι η συμφωνία, ε, της Συμφωνίας των Παρισίων με διαφάνεια στη δράση, λογοδοσία για τη δράση, ενημέρωση των εταίρων στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, όλα αυτά πρέπει να συμφωνηθούν στο τέλος του χρόνου στη Πολωνία. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη συζήτηση από την COP22 ε, στο Μαρόκο το 2016 ε, έχουν να ξανασυναντηθούν ε, άρα είχαν τα δύο χρόνια αυτά για να συζητήσουν τους τρόπους υλοποίησης της Συμφωνίας των Παρισίων, τα μέρη της λύσης, να καλέσουν την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει, σε εθνικό επίπεδο να δραστηριοποιηθούν διάφοροι Και ζητούμε ε, ένα εγχειρίδιο, όπως το λέμε, εγχειρίδιο των Παρισίων για την υλοποίηση. Από αυτό περιμένουμε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες συμμετέχοντες, ε, από τους συμμετέχοντες που θα έρθουν στην Πολωνία. Κάτι άλλο που ανησυχεί την κοινωνία των πολιτών και τους ε, μη κρατικού ε, φορείς είναι η αποφάση των μεγάλων ε, εταίρων πρέπει προς όφελος των νησιωτικών αλλά και των μικρότερων κρατών να περιοριστεί η αύξηση θερμοκρασίας των 1,5 βαθμό Κελσίου. αν δεν το καταφέρουμε αυτό θα έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων και καταστροφές φυσικές πολύ σημαντικές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι μεσαίοι και μεγάλοι παράγοντες ε, όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλοι ε, άλλα μέρη στη σύνοδο αυτήν να δραστηριοποιηθούν για να επιμείνουν να ε, υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Πρόκειται για τη λεγόμενη ε, για το λεγόμενο διάλογο της Ταλανόης, γιατί είχε ξεκινήσει πέρσι από τον πρόεδρο των ε, νήσων Φίτζη. Από αυτό περιμένουμε πολλά. Στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο υψηλέ φιλοδοξίες, να γίνει η συζήτηση πάντα συνδεδεμένη με την βιώσιμη ανάπτυξη για τον περιορισμό της θερμοκρασίας και κάτι ακόμη που θα ε, ήθελα να επισημάνω και να σας στήσω να φέρετε στη συζήτηση έχει να κάνει βέβαια με την οικονομική υποστήριξη που θα προσφέρουν τα μέρη που θα επιτρέψει και πιο υψηλές φιλοδοξίες στις χώρες εταίρους αλλά και τους τρόπους και τους μηχανισμούς προσαρμογής ε, ιδιαίτερα για τις, για τις λιγότερο αναπτυγμένες και τις μικρές νησιωτικές χώρες όπου θα είναι και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πολύ πιο σοβαρές. Έτσι λοιπόν το εγχειρίδιο και το κεφάλαιο του σε σχέση με την λογοδοσία στα δημοσιονομικά δηλαδή που πάντα είναι ένας πολύ, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι των διαπραγματεύσεων όπως θα είναι και φέτος οπωσδήποτε ξέρεις τι υπάρχουν ε, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία θα πρέπει δηλαδή να προσδιορίζει ποιος πληρώνει πόσα ποιος είναι ο παραλήπτης, ο αποδέκτης των ε, ε, κονδυλίων. Αλλά και πάλι εδώ μπορεί η Ένωση ως μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακή βοήθειας αλλά και χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή συνολικά να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή όπου μπορούν οι χώρες εταίροι να συναντηθούν και να συνομιλήσουν, να συνανοηθούν με τους αποδέκτες οι χορηγοί και οι αποδέκτες μαζί μπορούμε νομίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αποδεκτή, ικανοποιητική και κυρίως για τη χρηματοδότηση της ε, κλιματικής αλλαγής ε, για τις πιο φτωχές και εκτεθειμένες τους κινδύνους ε, αυτούς χώρες. Όχι μόνο για την κλιματική, αλλά και για τους στόχους της χιλιετίας. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό και για σας όπως ξέρω είναι η χρήση της γης το 1,5% που ξέρουμε ότι έχει καταγράψει στην έκθεσή της η διακυβερνητική διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή και θα παρουσιαστεί ε, το φθινόπωρο φέτος έχει να κάνει με το πώς μπορεί να περιοριστεί το σε 1,5 ε, βαθμούς Κελσίου ε, η αύξηση της θερμοκρασίας που σημαίνει για ορισμένες χώρες μέχρι και δύο βαθμούς συνολική αύξηση όπως ε, για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Βεβαίως ε, υπάρχει πολύ μεγάλη συνάφεια μεταξύ της αύξησης θερμοκρασίας και της χρήσης της γης, γιατί αναλόγως της χρήσης της γης μπορεί να περιοριστεί σημαντικά η ε, αύξηση της θερμοκρασίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε όρους ε, εκπομπών άνθρακα, σε όρους παραγωγής τροφίμων, σε όρους γεωργικής ε, παραγωγής, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα το κεφάλαιο χρήση γης. Και πρέπει να κοιτάξουμε και τις ε, βράχοι πρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες, αλλά και τις συνθήκες που προκύπτουν από τη φυσιολογική χρήση. Όπως είπα, πρόκειται για μια σύνοδο η οποία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία μετά το Παρίσι, Μπορεί να μην είναι το τελευταίο, οπωσδήποτε όχι, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και, και περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή παρουσία. Πάντοτε είναι πολύ σημαντικό γιατί πιέζει προ περισσότερε φιλοδοξίε στην ευρωπαϊκή πλευρά και σε αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή σα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Είμαι στη διάθεση σα φυσικά ε, για οποιασδήποτε περαιτέρω ερωτήσει. Η πρόεδρο ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μακλίν. Μπορώ να ακούσω τώρα τους ε, συναδέλφους. Με την κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αναφερθήκατε σε λύσεις που απορρέουν από την φύση, από τη φυσιολογική χρήση. Ιδιαίτερα ε, τονίσατε τη χρήση της γης. Εμείς θες κάναμε μια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας για τις συνέπειες της παραγωγής ε, κακάο, και καφέ, όχι μόνο στην εργασία των παιδιών, αλλά και στην αποψήλωση των δασών. με εκτιμήσεις ε, που δίνουν ένα 80% της αποψήλωσης ε, ως αποτέλεσμα της εκπέκτασης της γεωργικής παραγωγής. Ρωτώ λοιπόν τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το αποφύγουμε αυτό. Εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά την λύση της φυσιολογικής ε, ε, χρήσης, ε, ίσως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε κάποιες άλλες λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερο να επεκταθείτε στο θέμα της χρήσης της γης. Και επίσης ε, χρήση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Πώς εξετάζεται, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει. Ε, δεδομένου ότι μεγάλο κομμάτι της γεωργικής παραγωγής είναι τώρα η σόγια και το φινικέλαιο. Η COP24 πώς βλέπετε ότι θα χειριστεί τα θέματα αυτά. Ο κύριος Βέντα. Θα ήθελα κι εγώ να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. τη ευθύνε που αναφερθήκαν και νωρίτερα σε σχέση με του στόχου της χιλιετίας. Βεβαίως υπάρχουν τομεί οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους ε, και πάντως στις λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες υπάρχουν ζητήματα ζωτικής σημασίας. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα δηλαδή ο πληθυσμός μιας χώρας ε, από τις λιγότερο ανεπτυγμένε να προχωρήσει στη γεωργική του παραγωγή για να έχει επαρκή ε, ε, να έχει επάρκεια επιστημιστική. Επομένως, ε, μπορούμε βεβαίως με την ε, εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων αυτών να τους πούμε ότι πρέπει να προσέχουν πώς παράγουν και, να, και τι χρήση γης θα κάνουν, αλλά και αυτοί θα πρέπει να ζήσουν. Και άρα μπορεί αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα τελικά την καταστροφή της φύσης και του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Ωραία, Καλώς. Απαντήστε παρακαλώ. Θα προσπαθήσω, αλλά δεν είναι όλα αυτά δικιά μου αρμοδιότητα στην οργάνωσή μας. Πάντως από τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα για την προσαρμογή έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος και υπάρχουν πολλές προσπάθειες για προσαρμογή στην ε, Συμφωνία για το Κλίμα από πολλές ε, χώρες, ε, κοινότητες Προσπαθούμε να δούμε ακόμα και μικρές λύσεις, όχι πάντα μεγάλες υποδομές, αλλά συμφωνώ ότι είναι ένα ε, βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει και με την επέκταση της γεωργίας ε, και την ε, αναδάσωση. Προσπαθούμε να πετύχουμε τους βιώσιμους στόχους. Οπότε πρέπει να δούμε και τι είναι εφικτό και τι όχι. Σίγουρα να μην υπάρξει αποψήλωση των δασών, εννοείται ούτε να πηγαίνουν χρήματα για τέτοιου είδου προγράμματα. Αντίθετα, για προγράμματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ε, κίνητρα, ώστε να μην γίνεται αυτή η αποψήλωση, αλλά να βρεθούν άλλες λύσεις. Υπάρχει και η παγκόσμια διευκόλυνση για το περιβάλλον και τα πράσινα κονδύλια. Τώρα για τα βιοκαύσιμα, δυστυχώ δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν έχω ενημερωθεί. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι στην Oxfam και αλλού, στις μεταφορές. Έχουμε συναδέρφους που δουλεύουν για αυτά τα πράγματα και μπορώ να σας παραπέμψω σε αυτούς. Τώρα για τροφή και ασφάλεια, παραγωγή τροφίμων Σίγουρα εδώ έχουμε μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες και τα μέλη μας είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες και συζητούν με τους εταίρους μας εκεί για να βρεθούν καλές λύσεις. Πραγματικό όμως πιστεύω ότι από τα καλύτερα αποτελέσματα που είχαμε, κυρίως στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών, είναι μικρά προγράμματα Πρέπει να φτάσουμε σε τέρους, σε πολύ μικρές κοινότητες και προγράμματα, τα οποία από μόνο τους ίσως δεν μπορούν να σταθούν, αλλά προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία. Οπότε να κοιτάμε και προγράμματα που, χρησι... που χρηματοδοτούνται ίσως από κονδύλια διεθνή για το περιβάλλον κτλ. που όμως ε, δεν καταφέρουν να φτάσουν σε αυτά τα μικρά προγράμματα. Οπότε οι τοπικές κοινότητες, οι τοπικοί παράγοντες πρέπει να ενημερωθούν, να ξέρουν ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια. Είναι βασικό αυτό να το ξέρουν οι χώρες εταίροι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μακλίν για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστούμε και Ελπίζω να μπορείτε να μείνετε και άλλο εδώ μαζί μας. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα και θα συζητήσουμε... το ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, έτσι. Το αργότερο, την 3η 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, οι σκιώδεις συζητητές των ομάδων μπορούν να στείλουν προτάσεις για αλλαγές στο σχέδιο. Να τη στείλουν στη γραμματέα, στη γραμματεία που η οποία θα φροντίσει να φτάσουν αυτές οι προτάσεις στους άλλους και όδους αλλά και σε μένα και στην πρόεδρο εννοεί προφανώς η αντιπρόεδρος. Θα καταλήξουμε έτσι σε συμφωνία τελικά για ένα σχέδιο τροπολογιών. Οι συντονιστές μας στη συνέχεια θα εγκρίνουν το σχέδιο αυτό, το οποίο τελικά θα εγκριθεί και στην Επιτροπή μας. Έτσι λοιπόν, με καλό πνεύμα συνεργασίας από όλους, στις 29 και 30 Αυγούστου που θα συνεδριάσουμε εδώ θα μπορέσουμε και να τα εγκρίνουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να στείλουμε το σύνολο αυτό των τροπολογιών μας στην Επιτροπή ΕΝΒΗ έγκαιρα πριν να ψηφίσουν. Έτσι λοιπόν, επικεντρώμενες στις αρμοδιότητες της δικιάς μας Επιτροπής, αυξάνουμε τις πιθανότητες να συμπεριληφθούν οι τροπολογίες μας αυτές στο τελικό ψήφισμα της ΕΝΒΗ. Αυτά. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νίλς Σούστερ. Εσείς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλει βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύ σημαντική δουλειά σε αυτό το κρίσιμο ψήφισμα και ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη τη Επιτροπή ΔΕΒΕ για τα σχέδια τροπολογιών. Ευχαριστώ επίσης ε, την ε, φίλη από το δίκτυο κλιματικής δράσης που περιέγραψε πάρα πολύ καλά την κατάσταση, το πού βρισκόμαστε, πόσο σημαντικά είναι, σημαντικό είναι να επιτευχθούν ε, οι στόχοι και οι φιλοδοξίε για την COP24. Συμφωνώ σχεδόν σε όλα. Θα ήθελα απλώ να συμπληρώσω με την ανάλυση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί ω Επιτροπή βλέπουμε για το 2018 δύο προτεραιότητε. Καταρχά, την ολοκλήρωση του εγχειριδίου κανόνων τη COP24 με του κανόνε που είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία και από αυτή τη ενία θα έχει τεράστια σημασία η COP24 ως ε, επόμενο βήμα της COP21 ε, των Παρισίων. Το άλλο θέμα που επίσης αναφέρατε ε, και η σημασία είναι ότι καταγράφουμε την πρόοδο, τις προσπάθειες και τις περαιτέρω ανάγκες για προσπάθειες. Έτσι γίνεται μια απογραφή ε, ένα στιγμιότυπο της κατάστασης. Για το εγχειρίδιο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο, πλήρες, ε, ολοκληρωμένο, με θέματα που βεβαίως θα καλύπτουν και τον περιορισμό και την προσαρμογή. Και στην προσαρμογή βάζω βέβαια και την χρηματοδότηση για την ε, κλιματική αλλαγή. Θα επιτρέψει να μας δώσει περισσότερη ευελιξία στην προσαρμογή μας, ε, στην προσαρμογή των δυνατοτήτων, ε, τη δυνατότητα να επαληθεύεται η υλοποίηση από όλα τα μέρη των στόχων και ταυτόχρονα θα μας δώσει μια σαφή εικόνα για το που πρέπει να πάμε και σε αυτό πιστεύουμε ότι ένα πλαίσιο διαφάνειας ενισχυμένο με βάση το άρθρο 13 της ισχύουσας ε, συμφωνίας πλαισίου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη διαφάνεια. Θα θέλαμε μια μία δέσμη κανόνων ε, συμμόρφωσης ε, και επιβολής σε σχέση με τις προτάσεις αυτές, γιατί μπορεί να υπάρχουν οι κανόνες συμμόρφωσης, αλλά πρέπει να έχουν και κάποιες συνέπειες. Συγκεκριμένη στόχη. Ε, περιμένουμε από τις κυβερνήσεις ε, να αναλάβουν μετά την COP24 συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κατόπιν της, ε, του διαλόγου της Ταλανόης. Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται οπωσδήποτε και στο πλαίσιο της έκθεσης IPCC για, το 1, για τον 1,5 βαθμό Κελσίου μείωση περιμένουμε ε, αμέσως πριν από την Σύνοδο της Πολωνίας που επίσης θα είναι πολύ σημαντικό ε, βήμα. Στο διάλογο της Ταλανόης λοιπόν έχουμε προσπαθήσει να πούμε εμείς πώς βλέπουμε τα πράγματα και τι έχουμε κάνει, τη δική μας ιστορία που είναι μια ιστορία επιτυχίας γιατί καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο να, υλοποιήσουμε, να θέσουμε σε εφαρμογή όλα τα δεσμευτικά νομοθετήματα για την υλοποίηση των δικών μας, ε, του, ε, του δικού μας τμήματος των υποχρεώσεων. Άρα έχουμε κάνει αυτό που οφείλαμε. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε να αφηγηθούμε μια ιστορία και επιτυχίας αλλά και φιλοδοξιών και ο Επίτροπος οπωσδήποτε θέλει να ενισχύσει το επίπεδο φιλοδοξίας. Στην εκδήλωση λοιπόν που κάνουμε για το, είναι, για το διάλογο της Θαλανόης έχουμε, καλέσει, έχουμε προσκαλέσει εταίρους να έρθουν να μας πούνε τη δική τους ε, ιστορία, τις δικές τους ε, προτάσεις και ιδέες επίσης. 29 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει πάλι στη δεύτερη πολιτική φάση του διαλόγου της Θαλανόης. COP24. Η COP24 όμως δεν θα εξαντληθεί στην ε, Ταλανόη. Θα έχει και τεχνικούς κανόνες και θα αποτελέσει και μια λιδία λίθο της πολυμερού συνεργασίας. Πολύ σημαντική δοκιμασία για το εάν μπορούμε να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν έχουμε περιθώριο δηλαδή πιστεύω να αποτύχουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε. Πρέπει να φέρουμε εις πέρας όλες τις ε, προτάσεις για να προχωρήσουμε. Έχει βέβαια ηγετική θέση παγκοσμίω η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Με βάση και τις εξελίξεις που είδαμε πρόσφατα στη, στην πολυμερή τάξη πραγμάτων και του, την ομάδα των 7, την G7, αλλά και γενικά τις μεγάλες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δεδομένο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οργανώσει για τις 19 Ιουνίου την Υπουργική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή, τη λεγόμενη MOCA, Ministerial on Climate Action για την κλιματική δράση με την Κίνα και πολλούς άλλους εκπροσώπους 36 ε, κρατών μεγάλων οικονομιών σε μεγάλο βαθμό αλλά και των πλέον ευάλωτων ε, στην κλιματική αλλαγή κρατών. Η δεύτερη υπουργική μόκα είναι αυτή, η προηγούμενη ήταν πέρσι. Την οργανώνουμε και όσα απάντηση στις προθέσεις που έχουν ε, εκδηλώσει οι ΗΠΑ για αποχώρηση από τη Συμφωνία των Παρισίων. Ήταν μια απάντηση για να δείξουμε ότι υπάρχει ένα νέο φόρουμ μέσα από το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε και να ε, ε, αναπτύξουμε εταιρικέ σχέσεις με πολλές άλλες και σημαντικές χώρες του κόσμου. Πέραν της ΜΟΚΑ, ο Επίτροπος Κανιέτε έχει μιλήσει για μια πολιτική, συμφωνία πολύ σημαντική για την ενέργεια επί παραδείγματι, όπου έχουμε συμφωνήσει από το 27% των ανανεώσιμων να αυξήσουμε, 26-27% να αυξήσουμε σε 32 και 32,5% ε, τις φιλοδοξίες μας. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε και ο Επίτροπος, θα επιτρέψει αύξηση του στόχου μείωση των εκπομπών από, 40 έως 40, ε, από το 40% στο 45% ακόμα μέχρι το 2020 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη της ΚΑΠ 24 λοιπόν ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρόκειται για ανακοινώσεις σημαντικές, ανακοινώσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε την ε, ε, δυναμική ενόψη του Κατόβιτσε το Δεκέμβριο και βέβαια να βοηθήσουμε και όλους τους λοιπούς εταίρους που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την, ε, προς, τη στράτευση τους, τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις τους εν ώψη της ε, Συνόδου και πριν από την ΚΟΠ θα επιβεώσει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για μια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έως το 2020 ήδη έχουμε κάνει τις προτάσεις. Θα εξετάσουμε διαφορετικά σενάρια με μηδενικά, καθαρά μηδενικά αέρια του θερμοκηπίου έως το 2050. Αυτό είναι ένα σενάριο. Επίσης, Ε, θα στηριχθούμε στις ε, προτάσεις του πάνελ ε, για την κλιματική αλλαγή με το 1,5 με το 1,5 βαθμούς Κελσίου. Εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με όραμα, όχι τόσο με συγκεκριμένε προτάσεις από πλευρά της Επιτροπής, αλλά θα αναλύσουμε εννοείται τις προτάσεις και τις συζητήσεις όλες για περαιτέρω χρήση. Όλα αυτά για να ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουμε αυτές τις δύο μέρες μια πολύ σημαντική διάσκεψη των εμπλεκομένων περί τους χιλίους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες είχαμε αυτές τις δύο ημέρες στις Βρυξέλλες με μια δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική που θα δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο ε, για να συμμετάσχουν και διαγραμμικά οι ενδιαφερόμενοι για τις επόμενες 12 εβδομάδες και που τελικά θα δώσει αποτελέσματα με μία πρόταση τον Νοέμβριο. Για την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή, δύο λόγια επιτρέψτε μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να ε, συμβάλλει στο συλλογικό στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ω ως συλλογικό στόχο για τις, ε, για λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και προτείνει ω εκ τούτου ε, το τμήμα που αφορά την κλιματική αλλαγή στις ε, προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές να αυξηθεί από το 20% στο 25% χρηματοδότης για το κλίμα και βέβαια η αναπτυξιακή βοήθεια ε, χρησιμοποιεί πάντα την, τα αποθεματικά για να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μέτρα περιορισμού και μέτρα προσαρμογής σιγά σιγά με την αλλαγή της στάθμισης που έχουν μέσα στις πολιετήσεις νοσονομικές προοπτικές έρχονται σε ισότιμο ε, ποσοστό πλέον. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά εξασφαλίζοντας ασφάλεια για όλους τους ε, ενδιαφερομένους, για το κοινό, για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστούμε ιδιαίτερο το Κοινοβούλιο για τη συνεργασία και προσβλέπουμε βέβαια στη συνεργασία ενόψη της COP24 στο Κατόβιτσε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σούστερ. Έχουμε και έναν ακόμη ομιλητή από τη ΓΔ Τεύκο. Κογιέται. He's, he's not here. Δεν είναι εδώ. Ναι, κογιέται. όχι. Ε, δεν είναι εδώ. Ε, τον ε, αντικαθιστώ. Είμαι ο αρμόδιος Γενικός Διευθύντης της ΤΕΦΚΟ για την συνεργασία. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σχόλια σε σχέση με αυτά που είπαν οι ευρωβουλευτές πριν για την αντι... το πώς αντιμετωπίσουμε ε, την απερίμωση ε, και τα προβλήματα της γεωργίας. Σίγουρα είναι πολύπλοκα ζητήματα και οι συνθήκες διαβίωσης επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ε, για τον κόσμο ιδίως που ζει στην Ήπετρο όπως και ο κύριος Βέντα πολλοί έχουν κάποια δράση που δεν είναι και κάποια συμπεριφορά που δεν είναι ίσως περιβαλλοντικά υπεύθυνη ακριβώς λόγω των προβλημάτων. Εμείς προσπαθούμε ε, στην Κομισιόν να τα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Δεν μπορέσαμε σίγουρα να φτάσουμε σε κάθε απομακρυσμένη τοπική κοινωνία σε όλο τον κόσμο. Ε, Παρ' όλα αυτά έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ε, παγκόσμιας φύσης, όπως παραδείγματος χάρη Reducing Emission for ε, Deforestation, το RED όπως λέγεται, και έχουμε και μια συμμαχία, παγκόσμια συμμαχία για το κλίμα, Global Climate Alliance. Επίσης ε, Προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην προσαρμογή στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας και να στηρίξουμε τις κοινωνίες που πειράζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Φυσικά ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος είναι κάτι σημαντικό και υπάρχουν μέτρα που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο, ιδίως στις χώρες που έχουν έναν μεγάλο βιομηχανικό κλάδο αλλά όταν μιλάμε και για τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ε, εκεί ε, πρέπει να γίνει διαφορετική προσπάθεια. Αλλού πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Επίση, δίνουμε έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος τρόπος. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για να μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τις πολιτικές στις οποίες αναφερθήκαμε. Παραδείγματι, μέσα της ασοκομείας. Πώς να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, αν δεν υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης, ε, ε αν δεν υπάρχουν ε, και δασονόμοι, για να μην υπάρχει ε, εμπρισμοί παράνομοι ή να μην καίνε βιομάζα κάποιοι. Υπάρχει ένα πακέτο μέτρων για τις χώρες ΑΚΕ Είμαστε στη δεύτερη φάση της συμμαχία για το κλίμα, 70 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πενταετία. Είναι ο προπολογισμό και ξεκινούν προγράμματα σε διάφορες χώρες. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα, να έρθετε σε επαφή μαζί μα και θα σας δώσουμε τα χάρα πληροφορίες. Thank you very much. we... Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε όλους τους ομιλητές τώρα από την πλευρά της Κομισιόν. Δεν υπάρχει κάποιος βουλευτής που να θέλει να σχολιάσει, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό της μέσης διάταξης. Τέλη Αυγούστου ή ε, αρχές Σεπτεμβρίου θα ξανασυζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Αλλά προς το παρόν ολοκληρώθηκε η συζήτηση και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. που είναι η ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη. Μειώνοντας τη φτώχεια μέσω της τεχνολογίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων το Μάιο. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε το ζήτημα. Όλοι γνωρίζουμε πως η ψηφιοποίηση μεταβάλλει άρδιν τις κοινωνίες μας. Βέβαια, όπως είναι προφανές, είναι αυτή η επανάσταση δεν αποκλεί τις χώρες που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα. Στις αναπτυγμένες χώρες, στις ανεψόμενες χώρες σήμερα υπάρχουν Περισσότερα νοικοκυριά που έχουν κινητό τηλέφωνο από όσα έχουν πρόσβαση σε ρεύμα ή πόσιμο νερό, καθαρό νερό. Σίγουρα την ανάπτυξη αυτή την προκαλούν πιο πολύ τεχνολογικές αλλαγές, τεχνολογική πρόοδος, η ζήτηση και εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένε πολιτικέ. Ορισμένε από τι πιο μεγάλε προκλήσει που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τα πολέμηση του ψηφιακού χάσματο. Αυτό το ψηφιακό χάσμα προκαλείται από διαφορές ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα, ε, την προστότητα των τιμών ε, ή τον ψηφιακό εγγραμματισμό ή αλφαβητισμό. Επομένως χρειάζονται καλές πολιτικές που θα εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία των ψηφιακών υποδομών και θα βελτιστοποιήσουν, θα μέγιστοποιήσουν τα κοινωνικά, οικονομικά και δημοκρατικά ωφέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επίσης τα κράτη-μέλη και άλλοι ε, χρηματοδότες, δωρητές ήδη στηρίζουν την ψηφιοποίηση και στα τελευταία 20 χρόνια και η Κομισιόν υποστήριξε έργα στον τομέα αυτών, το ψηφιακό, συγκεκριμένα για την τελευταία δεκαετία, σε ψηφιακές πρωτοβουλίες διατέθηκαν περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο είναι σημαντικό η προσέγγιση της Κομισιόν Digital for Development d να μην εφαρμοστεί απομονωμένα, αλλά να ενταχθεί στις ε, αναπτυξιακές στρατηγικές συνολικά, αλλά και στον διάλογο με τις χώρες εταίρους για θέματα πολιτικής. Και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, καταρχάς ε, με τον εισηγητή μας, ε, Μπρόγκταν Μπρούνον Βέντα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά την στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πέρυσι να εκπονήσει έκθεση. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέρφους και βέβαια από τη γραμματεία το προσωπικό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ψηφιοποίηση στην ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να μειωθεί η φτώχεια, γιατί δημιουργεί νέε ε, δυνατότητες απασχόλησης. Η Αφρική και η Λατινική Αμερική δυστυχώς έχουν μείνει πολύ πίσω και χάνουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν ε, τις ε, δυνατότητες να πετύχουν τους βιώσιμους στόχους, τους στόχους της χιλιετίας. Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές για την ψηφιοποίηση, αυτό λέω στο πρώτο μου τμήμα και στο δεύτερο τμήμα αναφέρω τους διάφορους τομείς που έχουν να κάνουν με το φαινόμενο αυτό. Δουλεύοντας για την έκθεση αυτή, οργανώσαμε ακρόαση, είχαμε διαβουλεύσει, συζητήσαμε με τους ενδιαφερόμενους από όλες τις πλευρές και για δύο μέρες μαζί με τη γραμματεία οργανώσαμε και μία συνάντηση multi-stakeholders όπου συζητήσαμε το σχέδιο γράφου. Υπήρχε μάλιστα και το αίτημα από τους σοσιαλιστές, από τον κύριο Γκερέρο Σαλόμ που είναι σκιώδης ε, εισηγητής, να προσθέσουμε κάτι για την ανθρωπιστική αρρωγή στο σημείο 20. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία fast track. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στο τέλος του καλοκαιριού 31 Αυγούστου είναι η προθεσμή για την υποβολή τροπολογιών. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και για τις τροπολογίες 24 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 9 Οκτωβρίου. Οπότε προσβλέπω τα σχόλιά σας και θα δω βέβαια και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε εδώ κανένα σκιώδη Α, έχουμε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Που μόλις, μόλις έφτασε. Φλόρενς Μακτέλερη, από τους πράσινου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τόσα μας είπε για ένα πρώτο σχέδιο. Έχω να κάνω κάποια σχόλια για την πρόταση αυτή. Πέρα από τις γενικότερες προσπάθειες για την αναγκαιότητα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτήν την ε, άποψη για την τεχνολογία, αυτό το όραμα, ώστε να φτάσει και στον Νότο. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε και πιο επικριτικοί όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών και πώς φτάνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κάτι το οποίο λείπει κατά τη γνώμη μου και ως πράσινη θα υποβάλουμε σχετικές προτάσεις. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τις προτεραιότητές μας για την ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες οι ανάγκες δεν είναι τόσο πολύ μεγαλύτερη ψηφιοποίηση, εντάξει χρειάζεται και αυτό, αλλά περισσότερο χρειάζεται βασική εκπαίδευση, βασική υγεία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι δεδομένου ότι ο προπολογισμό είναι περιορισμένο, πιο πολύ πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπιστούν αυτέ οι βασικέ ανάγκε και μετά να περάσουμε στην ψηφιοποίηση. Κυρίω σε χώρε οι οποίε βρίσκονται σε διαδικασία βιομηχανοποίηση. Ε, τα πλαίσια δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Οπότε θα έλεγα να ε, δούμε λιγάκι πώς θα θέσουμε τις προτεραιότητές μας, μέσα σε ένα περιορισμένο προπολογισμό φυσικά. Έπειτα πρέπει να δούμε το ψηφιακό χάσμα. Οι προτάσεις που κάνουμε πρέπει να φροντίσουμε να μην αυξάνουν το ψηφιακό χάσμα. Παράδειγμα, Γεωργία. Γνωρίζουμε καλά ότι η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογίες μπορούν να στηρίξουν ένα σύστημα ή ένα άλλο. Σε πολλές χώρες όμως βλέπουμε ότι είναι η βιομηχανία τροφίμων που υποφελείται τελικά από τις νέες ε, τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση. Και ελπίζω ότι και στο Νότο θα μπορέσουμε την ψηφιοποίηση να την θέσουμε στην υπηρεσία της ε, αγροοικολογίας που όπως λέει και ο ΦΑΟ είναι το σύστημα του μέλλοντος για να μπορέσουμε να έχουμε αρκετά τρόφιμα για τον κόσμο. Κάτι άλλο. Δημοκρατία και ασφάλεια. Και εδώ έχουμε πολλούς στόχους, κυρίως για την ασφάλεια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με την ε, αύξηση των νέων τεχνολογιών, στις επικοινωνίες κτλ. Έχουμε και μια αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίως σε αυτές τις χώρες του Νότου, όπου η ρύθμιση, οι θεσμοί είναι πολύ πιο αδύναμοι από ό,τι στις χώρες μας. Οπότε νομίζω ότι και αυτό πρέπει να σημειωθεί στην έκθεση και να προσθεθεί στον προβληματισμό. Κάτι άλλο το οποίο νομίζω δεν υπάρχει στην έκθεση, δεν είδα, είναι οι οικολογικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών. Ξέρουμε ότι το οικολογικό αποτύπωμα είναι πολύ μεγάλο των νέων τεχνολογιών το cloud που λέμε, το νέφος το ηλεκτρονικό που νομίζουμε ότι είναι άϊλο, δεν είναι άϊλο. Αυτό σημαίνει δορυφόρη, σημαίνει κατανάλωση ενέργειας κλπ. κλπ. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ψηφιοποίηση του κόσμου ολόκληρου σε βάρος της οικολογικής διάστασης και του πλανήτη. Και έπειτα για τη χρηματοδότηση. Πρέπει να δούμε πώς θα συνδυάσουμε την ε, ψηφιακή διάσταση με τις οικονομικές ικανότητες των χωρών. Αυτά είναι τα διάφορα σημεία που ήθελα να προσθέσω. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε πάρα πολύ καλά να συνεργαστούμε για αυτά τα σημεία που πιστεύω ότι είναι πολύ βασικά για να βελτιωθεί το σχέδιο έκθεσης και να πετύχουμε τους στόχους ε, που έχουμε για την ψηφιοποίηση των χωρών του Νότου. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ωραία, τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παόλο Τσικορέλη, σωστά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ονομάζομαι Πάολο Τσικαρέλη. Στην ΤΕΦΚΟ, αναπτυξιακή συνεργασία, με αρχής ψηφιοποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την επιτροπή σας που άνοιξε το θέμα αυτό προς συζήτηση. Είναι ένα θέμα που αναφύεται τώρα στην, στο θεματολόγιο μας, στο πρόγραμμά μας. Μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισκύπτει στο θέμα αυτό. Ήδη η Επιτροπή σας μας επέτρεψε να παρουσιάσουμε το έργο μας την ψηφιοποίηση. Το έγγραφο εργασία απευθύνεται στο προσωπικό για την ψηφιοποίηση στην ανάπτυξη και τη στρατηγική προσέγγιση που αναπτύσσεται μέσα από αυτό το έγγραφο εργασία που απευθύνεται στο προσωπικό. Με την ε, σημερινή συνάντηση νομίζω μπορώ να σας ενημερώσω για, την, ε, για τις τελευταίες προόδους, τι έχουμε καταφέρει, τι κάνουμε από την εποχή που ξεκίνησε αυτό το έγγραφο εργασίας για το προσωπικό. 300 και 350 εκατομμύρια για την ψηφιοποίηση έχουμε αφιερώσει τελευταία δεκαετία ε, και θα ήθελα συγκεκριμένα για το 2017 να σας δώσω στοιχεία 110 και εκατομμύρια για τις υποδομές της ψηφιοποίησης και την ψηφιακή συνδεσιμότητα. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 300 εκατομμύρια που είχαμε για τη δεκαετία του 6 έως 16. Και όπως βλέπετε έχουν αυξηθεί οι ρυθμοί υποστήριξη τη ψηφιοποίηση. Όπω είπα, πρόκειται για ένα έγγραφο εργασία απευθυνόμενο στο προσωπικό, στο οποίο η ψηφιοποίηση περιγράφεται, χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αναπτυξιακής μας συνεργασίας. Δεν τη βλέπουμε σαν ένα ξεχωριστό τομέα, δηλαδή την ψηφιοποίηση και για να αναφερθώ στα όσα είπε η συνάδελφος νωρίτερα, θα ήθελα ε, να, σας να ότι δεν μιλούμε για ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των προτεραιοτήτων, υγεία, η ψηφιοποίηση, η εκπαίδευση, η ψηφιοποίηση. Όχι, κοιτούμε να δούμε πώς μπορούμε με την ενίσχυση της ψηφιοποίησης μπορούμε να στηρίξουμε αποτελεσματικά ουσιαστικά το τομέα της εκπαίδευσης, το τομέα της υγείας, το τομέα της γεωργίας. Άρα δεν, δεν πρέπει να αναζητεί κανείς τις προτεραιότητες. Απλώς αντιλαμβανόμαστε ότι μέσω της ψηφιοποίησης μπορούμε να ενισχύσουμε όλους τους πρωτογενείς μας στόχους. Και όταν μιλώ για ψηφιοποίηση, Επαραδειγματι ε, στο τομέα της υγείας, ε, η συζήτηση για την ψηφιοποίηση ξεκινάει πάντα από την αφετηρία της υγείας. Δηλαδή, κοιτούμε να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε την υγεία με εμπειρογνώμονες της υγείας, και προσπαθούμε μέσα σε αυτό να δούμε η ψηφιοποίηση πώς μπορεί να συμπληρώσει και να υποστηρίξει την πολιτική για τη δημοσία υγεία. Άρα δεν υπάρχει όπως πανταγωνιστική σχέση, αλλά ε, τρόπος ενίσχυσης της αναπτυξιακής μας συνεργασίας. Το ίδιο και στην ενέργεια. Υπάρχει σαφή συνάφεια μεταξύ ψηφιοποίησης και ενέργειας. Και η ψηφιοποίηση μπορεί οπωσδήποτε να ενισχύσει τα συστήματα προμήθειας ενέργειας. Και βλέπουμε στην Αφρική πολύ συχνά ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να έχει ένα ψηφιακό εργαλείο, μηχάνημα, ένα smartphone και με τον ίδιο τρόπο προσπαθεί να εξασφαλίσει ο κόσμος και ανανεώσιμες ε, πηγές ώστε να μπορούν να ε, φορτίζουν τα smartphone ή όποιο άλλο ε, μηχάνημα επικοινωνίας έχουν. Θέλουν παραδείγματι ηλια... Ε, θέλουν παραδείγματι power bank με ηλιακές κυψέλες. Τώρα για να προχωρήσω στη χρηματοδότηση ψηφιακής, ε, των ψηφιακών οικοδομών. Πέραν αυτών που σας ανέφερα νωρίτερα, έχουμε επενδύσει 200 εκατομμύρια για προγράμματα που υποστηρίζουν τους τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, ε, της γεωργίας και της δημόσιας υγείας. Και επίσης από την έκθεση της Επιτροπής σας βλέπουμε ικανοποίηση την αναφορά στην ε, ανοιχτή προσέγγιση, μια προσέγγιση που δεν θα αποκλείει κανέναν. Εξετάζοντας λοιπόν αυτό το θέμα της κάλυψης ε, της ψηφιακής αναφερόμαστε, έχουμε μια ιδιαίτερη μνήα με ένα πρόγραμμα 38 εκατομμυρίων στους πιο φτωχούς και στις γυναίκες, ειδικά αλλά ταυτόχρονα ετοιμάζουμε και κάποιες μελέτες μέσα από τις οποίες θα εξετάσουμε πώς μπορούμε καλύτερα να στηρίξουμε τις γυναίκες και τις δυνατότητές τους για αυτόνομη δράση μέσα από ένα ε, κομμάτι, ένα κεφάλαιο ψηφιοποίησης στα προγράμματά μας. Κοιτάμε και τον ιδιωτικό τομέα οπωσδήποτε, γιατί και αυτός έχει πολύ σημαντικό ρόλο να μιλούμε για την ψηφιοποίηση. Πρόκειται για εταίρο κρίσιμη σημασία όταν μιλούμε για την ε, απελευθέρωση του δυναμικού της ε, ψηφιακής οικονομίας. Και σε αυτό έχουμε διάφορα παράθυρα ανοίξει, εκ των οποίων το ένα αφορά συγκεκριμένα την ψηφιοποίηση, που έχει δεχτεί πολλές προτάσεις. Και έτσι από τις δύο προτάσεις που έχουμε ε, ετοιμάσει και πάνε για κλείσιμο. Η μία αναφέρεται στην ψηφιακή δημόσια υγεία και η άλλη στην ψηφιακή οικονομία. Αυτά κλείνοντα, θα θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες προς τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής σας. Η υλοποίηση των αρχών της ψηφιακής ανάπτυξης ε, σε τις προτάσεις νομίζω μόνο κέρδος μπορεί να φέρει. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος ε, από την Επιτροπή ή από τους βουλευτές. Κύριος ε, Μαξιρίνη. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο για κάτι που είπε ο ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον οικολογικό αντίκτυπο. Πρέπει να εμβαθύνεται λίγο παραπάνω, διότι είχαμε την ε, συζήτηση για τα ενεργειακά ζητήματα, ενεργειακή απόδοση κτηρίων, ε, αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Τα γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα αυτά. Δεν έχει, σταματή, δεν έχει ολοκληρώσει ε, τον προβληματισμό τη Κομισιόν για τον οικολογικό αντίκτυπο που θα έχουν οι τεχνολογίε. τεχνολογίες. Φυσικά και οι νέε τεχνολογίε μπορούν να συνεισφέρουν στη διαχείριση, το smart grid, τα εφή δίκτυα κτλ. Ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που θα χρησιμοποιούν περισσότερο. Αλλά αυτά εδώ που έχω στο χέρι μου έχουν έναν αντίκτυπο υλικό. Δεν είναι κάτι άλλο. Υπάρχει πρίζα ε, στην οποία μπαίνει ο φορτιστής ε, και αυτό, ε, όλα τα στοιχεία αυτά τελικά πηγαίνουν και μέσα σε ένα σε μια δεξαμενή αποδίκευση δεδομένω. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα που μπορούμε, θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στις μελέτες μας. Αυτό δεν γίνεται όμως μπορούμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση χωρίς μπούμεραγκ ε, γιατί πολλές φορές χάνουμε ε, σε ό,τι αφορά τον οικολογικό αντίκτυπο ή τη χρήση των πρώτων υλών. Δηλαδή ε, πρέπει να το δείτε ολιστικά το θέμα, γιατί δεν ισχύει πάντοτε ότι όλοι είναι κερδισμένοι, ότι είναι win-win και για όλες τις πλευρές. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη κάποια στιγμή και αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θέλετε να απαντήσετε. Συμφωνώ, αυτή είναι η απάντησή μου. Φυσικά και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το βλέπω πολύ θετικά. Και όσο προχωρούμε στην ανάλυση μας, σίγουρα θα το λάβουμε υπόψη το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο συγητής μας, ο κύριος Σεβέντα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να τα πω ισπανικά, αφού μόνο ένας και είναι εδώ, άρα μπορούμε να τα λέμε ισπανικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα σχόλιά σας σε σχέση με κάτι που είπες, συγγνώμη που σου μιλάω στον ελληνικό, ε, έχουμε το σημείο 13 για την ασφάλεια που λέω ότι είναι σημαντικό. Συμφωνώ ότι πρέπει να τα συνδυάσουμε. Ο ψηφιακό κόσμο ε, μπορεί να παρουσιάσει και κάποιου κινδύνου σε ό,τι αφορά τη Γεωργία το 18. Ναι, και για αυτά συζητούμε. Μιλάμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει στην έκθεση, έτσι, καταρχάς. Αυτό με το 20, την πρόταση του Ενρίκε Γκερέρο, το, με, ε, το έχω ήδη αναφέρει και η διακυβέρνηση είναι, είναι στο 22 σημείο. Επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να δούμε ε, και ποια είναι η δική μας προοπτική, αλλά και το τι ισχύει στις χώρες αυτές. Ε, υγεία, ε, υγιεινή, πράγματι, υπάρχουν, το είδαμε στις επαφέ μας, υπάρχουν χώρες στις οποίες όταν έχουμε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή, υπάρχουν κάποια σύγχρονα εργαλεία συγκέντρωση δεδομένων για τον ιό του έμπολα, για παράδειγμα υπάρχουν προβλήματα, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά και να προλάβουμε κάποιε καταστάσεις. Όπως και αν έχει, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μιλήσαμε πριν για την οικολογία και το κλίμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει και να προστατεύσουμε. Και θέλουμε να δούμε τι θέλουν αυτές οι χώρες. Αν έχουν να αντιμετωπίσουν επιδημίες ή το λοιμό, τον υποσυτισμό, άλλα προβλήματα. Δεν έχουν πρόσβαση. Επομένως, η αξιοποίηση της ψυχικής τεχνολογίας ε, μπορεί να βοηθήσει ίσως πιο γρήγορα, πιο εύκολα να φτάσουμε ε, σε αυτά τα... να πετύχουμε τους στόχους αυτούς της ε, βιώσιμης ανάπτυξης που θέλουμε. Φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ μας Περιμένω βέβαια και τις τροπολογίες που θα μου στείλετε και φαντάζομαι θα βελτιώσουν το κείμενο, αλλά ε, το λέω από τώρα ότι ήδη περιλαμβάνει το κείμενο μου κάποια από αυτά που είπατε. Μπορώ να εμβαθύνω περισσότερο για να μην ξεχάσουμε κάποια από αυτά τα οποία αναφέρετε. Πάντως ε, πνεύμα συνεργασία ε, υπάρχει από πλευρά μου και θα δούμε και τι τροπολογίε θα καταθέσετε εσεί, οι υπόλοιποι και θα βρούμε λύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βέντα. Ωραία. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 31η Αυγούστου στις 10. Εντάξει. Ωραία. Οπότε έληξε το θέμα αυτό. Για ώρα ερωτήσεων δεν έχουμε ερωτήσει. Εντάξει, αυτά. Σημείο 16. Διάφορα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα τον Αύγουστο, 29 Αυγούστου. Οπότε ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής μας και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Ελπίζω να έχουμε όλοι ένα όμορφο και ζεστό καλοκαίρι, όπου και αν βρίσκεστε και όπου και αν κάνετε διακοπές. Θα τα ξαναπούμε τον Αύγουστο.